Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Είμαστε λοιπόν η Επιτροπή ΕΜΒΗ για τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Είναι μεγάλη χαρά μου που έχω την τιμή να αναλάβω την Προεδρία τούτης της Επιτροπής. Θα ξεκινήσω με το πρώτο σημείο που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε χωρίς τροποποιήσεις το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν. Εγκρίνεται. Περνάμε μετά στις ανακοινώσεις της Προεδρίας. Ο Στεφάν Ντονέα αποτελεί πλέον τμήμα της γραμματείας ΕΜΒΗ από την 1η Απριλίου. Η Νόρα Κοβάτσεβα επανήλθε στην γραμματεία της Ένεβη μετά από ένα χρόνο ε, στην ε, Επιτροπή ΕΜΙΣ, οπότε είναι μαζί μας και πάλι από τις 10 Απριλίου. Καλωσορίζω και τους δύο εκ μέρους Επιτροπής ΕΝΒΗ. Θα περάσω μετά στις ανακοινώσει σε σχέση με τις συστάσει των συντονιστών από την 11η Απριλίου του 2017. Να σας πω πως σα έχουν μοιραστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε και εδώ πως εγκρίνονται. Δεν έχουμε αντίρρηση λοιπόν. Ε, από ό,τι βλέπω εγκρίνονται. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για τα πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια των ανθρωπίνων οργάνων ε, που χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις. Θα δώσω το ρόλο τώρα στον ε, κύριο Νίκελ Σνίκελς, με συγχωρείτε, που είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να κάνει μια σύντομη παρουσίαση ε, της εφαρμογής της οδηγίας αυτής που είναι η 53 του 2010, που είναι μια πετυχημένη, ένα success story της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσω με κάποια αριθμητικά στοιχεία. Το 2015 πάνω από 10.000 δωρήσεις οργάνων έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα πάνω από 33.000 μεταμοσχεύσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αύξηση της τάξης του 29% από το 2006, στοιχείο εντυπωσιακό. Η αύξηση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας βασικής αύξησης των ε, ζώων των μεταμοσχεύτων συν 56% και στους ε, αποθανόντες που δορίζουν μεταμοσχεύσεις η αύξηση είναι 21%. Δεν είναι μόνο εντυπωσιακό, αλλά είναι το καλύτερο νέο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους ασθενείς, μία και καταρχήν αποτελούν μονόδρομο και βεβαίως σώζουν ζωές. Δεν θα πρέπει όμως να επαναπαυθούμε. Δυστυχώς υπερβολικά πολλοί άνθρωποι περιμένουν όσο είναι στη λίστα αναμονής, όσο περνάνε τα χρόνια και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε συνέχεια. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποια άλλα στοιχεία που είναι οι δωρητές ανακράτως. θα δούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη. Μπορούμε όμως να δούμε πως ακόμα υπάρχουν βασικές ε, αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών στην Ισπανία και στην Κροατία έχουμε ένα εκατομμύριο ε, κατ' 40 δωρητές, που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά σε όλο το χρόνο. Με διαφορά τα όσα γίνονται σε άλλα κράτη-μέλη που μπορεί να έχουν και 10 φορές λιγότερες ε, ε, δωρήσεις οργάνων. Και μπορώ να σας πω πως οι διαφορές αυτές είναι και για τους εν ζωή ε, δωρητές, όπου στην πρώτη θέση βρίσκονται οι κατοχώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι τα στοιχεία μας οδηγούν στο μοναδικό συμπέρασμα που υπάρχει τεράστιο δυναμικό για περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να διδαχθούμε α, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, όπως η Κροατία διδάχθηκε από την Ισπανία και νομίζω ότι εκεί έχουμε επικεντρώσει και τις προσπάθειές μας τα τελευταία χρόνια για τα, μεταμοσχέσεις και την, τους δωρητές οργάνων έχουμε βασιστεί σε δύο σημεία. Έχουμε ε, την οδηγία του 2010, ένας πυλώνας που είναι τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας ε, για τους δωρητές οργάνων και τις μεταμοσχέσεις και την εθελούσια συνεργασία βασισμένη σε ένα σχέδιο δράσης που στηρίζει τις εθνικές αρχές και στους κλάδους που δεν καλύπτει η νομοθεσία, δηλαδή ε, την αποτελεσματικότητα του συστήματος ε, μεταμοσχεύσεων και την αυξημένη ε, προσφορά οργάνων. Ο λόγος για τον οποίο καλέσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα είναι η πρόσφατη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης για το πώς πάει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Πρέπει να σας πω πως ε, ε, είχαμε εισάγει μες οδηγίες αυτής τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας που καλύπτουν όλη την αλυσίδα ε, τροφοδοσίας, δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται η δωρεά μέχρι τη μεταμόσχευση και καλύπτουμε και όλα τα διάμεσα στάδια, ε, δηλαδή τη μεταφορά κτλ. Και αρχικά εστιάζουμε στο κατά πόσο υπάρχει η απαραίτητη εποπτεία του κλάδου από τα κράτη-μέλη. Και εδώ τα νέα είναι καλά. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ευδοδιγραμμιστεί με την οδηγία και έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες αρχές. Όμως, είναι διαφορετικά τα μοντέλα που χρησιμοποιούν για να καλύψουν την υποχρέωση εποπτείας. Άλλοι έχουν μία αρχή, άλλοι έχουν μέχρι τέσσερις. Από τη δική μας προπτική οπτική γωνία αυτό είναι απολύτως αποδεκτό, αρκεί οι κανόνες να είναι σεφείς, να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο το οποίο παρακολουθήσαμε ε, κατά τη διάρκεια αυτής της εφαρμοστικής διαδικασίας είναι τι γίνεται ε, με την απόκτηση οργάνων ε, από ιατρικές ομάδες άλλων κρατών μελών. Ε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και είναι ευκταίο γιατί δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη ένα κέντρο μεταμόσχευση πνευμόνων ή καρδιά. Είναι πολύ ακριβά τα προγράμματα αυτά. Δεν είναι αρκετέ ενδεχομένω οι μεταμοσχεύσει. Οπότε τα κράτη-μέλη συνάπτουν πολυμερεί ή διμερεί συμβάσει που τους επιτρέπουν να ε, χρησιμοποιήσουν την πραγματογνωμοσύνη των πιο έμπειρων χωρών για να ε, αποκτήσουν όργανα στις, ε, και να τα χρησιμοποιήσουν στις χώρες όπου υπάρχουν, υπάρχει λιγότερη εμπειρία. Και βέβαια αυτό λειτουργεί και αντίστροφα με αποτέλεσμα να συλλέγονται περισσότερα όργανα προς όφελος των ασθενών. Αυτή είναι η πραγματική ευρωπαϊκή συνεργασία βασιζόμενη στην αλληλεγγύη, στην πρόοδο και στα αποτελέσματα της εξαιρετικής δουλειάς που κάνατε και εσείς ε, για την οδηγία αυτή. Για το σχέδιο δράσης να σας πω πως εμείς χρηματοδοτούμε και project και μελέτες και σχέδια που επιτρέπουν συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Δηλαδή, να σας πω κάποια ε, παραδείγματα. Έχουμε προγράμματα αδελφοποίηση όπου οι πιο έμπειρες χώρε εκπαιδεύουν τους ε, λιγότερο έμπειρες. Επίσης ε, ε, εκπαιδεύουν τους συντονιστές μεταμοσχεύτεων και έχουμε και μία επικοινωνία όπου μπορούν μέσω αυτής της πλατφόρμας, της επικοινωνικής πλατφόρμας να χρησιμοποιούνται όργανα που έχουν δωρηθεί από αλλού και κυρίως για τα όργανα που χρησιμοποιούνται για παιδιά, μια και εκεί οι ιατρικές ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένε και ε, τα αποθέματα πολύ πιο περιορισμένα. Έχουμε και μια εργαλειοθήκη που επιτρέπει τις, πιο, ε, τις λιγότερο έμπειρε χώρε να αποκτήσουν τέτοια προγράμματα. Το σχέδιο δράσης έληξε το 2015 και αυτή τη στιγμή αξιολογείται και η τελική έκθεση θα σας δοθεί πριν το καλοκαίρι. Πρόσφατα λάβαμε και πολύ υψηλή χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ευγνωμόνες. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο μεγάλα ε, ε, έργα. Το ένα για τις ε, χρόνιες παθήσεις και το άλλο για την αύξηση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Εάν δεν έχετε αρκετά επιχειρήματα για να στηρίξετε την ευρωπαϊκή συνεργασία ε, στο κλάδο των, ε, της δωρεάς οργάνων και των ε, μεταμοσχεύσεων, να σας δώσω εγώ ένα επιχείρημα. Όχι μόνο σώζουν ζωές, αλλά έτσι εξοικονομείτε και πόρους. Και θα σας δώσω τα παραδείγματα που έχουμε στη διαφάνεια, που είναι παλιά στοιχεία, αλλά ε, παρόλα αυτά ισχύουν ακόμα αν αντί να κάνετε, διάλυ... Ε, αντί να κάνετε μοκάθαρση ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, κάνετε μεταμόσχευση νεφρού, μπορείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο να εξοικονομήσετε 80% των εξόδων για κάθε έτος ζωής. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια λίρες σημαίνει αυτό. Με καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή και την δυνατότητα ασθενής να επιτρέψει και στον εργασιακό βίο. Κλείνει λοιπόν έτσι η σύντομη παρουσίασή μου και θα ήθελα και μια φορά ακόμα να σα ευχαριστήσω, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που κάνετε στη δωρεά όργανων, στι μεταμοσχεύσει. Νομίζω ότι είναι η πραγματική, το πραγματικό success story τη Ευρώπη. Και εντάξει, καμιά φορά δεν είναι τόσο το γνωστό, συμβαίνει και με άλλες επιτυχίες της Ευρώπης. Εάν έχετε ερωτήσεις, οι συνάδελφοι και εγώ με μεγάλη χαρά να απαντήσουμε. Merci, merci beaucoup, euh, monsieur, monsieur le chef d'unité. Je rappelle que... Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δευθυντά, είσαστε, στην ΔΕΛΤΑ 4, ευθυντής. Θα δώσω τώρα στο λόγο, το λόγο στους συναδέλφους μας. Η κυρία Μέσμερ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την έκθεση την οποία παρακολούθησα πολύ προσεκτικά. Ήμουν και βουλευτή στην Βουλή της Κάτω Σαξονίας και γνωρίζω το πρόβλημα των δωρητών είναι πάντα μεγάλο, δεν υπάρχουν αρκετοί δωρητέ και απογοητεύτηκα λίγο για το ότι η Γερμανία δεν συνεργάζεται καθόλου. Ξέρω ότι έχουμε δυσκολίε. γι' αυτό το ερώτημα είναι πώ λειτουργεί το πράγμα. Λέτε ότι έχετε την οδηγία αλλά βεβαίως ε, είναι κάτι το εθελοντικό η συνεργασία των χωρών. Υπάρχει κάποια ανταλλαγή με συμμετοχή όλων των ε, χωρών. Συμμετέχουν και τα 28 κρατημέλη Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι απόρρισα με την συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί καλά η συνεργασία. Αφενός έχουν ειδικέ πτήσει. δεν ξέρω. Ε, δηλαδή εγώ θα σκεφτόμουν κάτι το πιο λογικό. Γειτονικέ χώρες, δηλαδή Κύπρος, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κάπως απομακρυσμένε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουν ή λειτουργούν όλα χωρίς πρόβλημα. Το δεύτερο ερώτημα και το τρίτο. Επειδή είπατε πως μια περίπτωση είναι η κάτω χώρες ε, μπροστά. Μα αν έχω ενημερωθεί σωστά, όταν ε, κάποιος εκεί πέρα υποκύψει, αυτομάτως θεωρείται ε, δωρητής, εκτός αν έχει δηλώσει το αντίθετο. Έχετε κάποια στοιχεία για το πόσες χώρες έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Γνωρίζω ότι στη Γερμανία δεν ισχύει αυτό και έχουν εντύπωση ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχουν νομίζω περισσότερα όργανα που δορίζονται. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταλή έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Επιτροπή. Θετικό είναι αυτή η αύξηση στα ποσοστά των δωρητών και το 29% που ακούσαμε είναι όμως ακόμα ανησυχητικό το ότι η ζήτηση για όργανα υπερβαίνει την προσφορά, όπως μας είπε ο εκπροσωπός της Κομισιόν στην παρουσίαση. Και είδαμε ότι πολλά άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ένωση, ενώ βρισκόταν αναμονή δωρητή. Και στο τέλος του έτους συνεχίζει να είναι Ανησυχητικό το ότι έχουμε 64.000 ασθενείς που παραμένουν σε λίστες αναμονής. Αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάγκη για να ασκήσουμε πίεση και να προωθήσουμε τον δωρεά οργάνων με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Και πρώτα θα ήθελα να υποφελθώ σε ευκαιρία για να τονίσω τη σημασία γενικότερα της δέωσης των οργάνων και υπάρχει το δίκτυο δωρεάς οργάνων όπου αναφέρεται τέλο πάντων ότι χωρίς τη δωρεά δεν υπάρχει ελπίδα. Όταν όμως υπάρχει δωρεά οργάνου υπάρχει επανάκαμψη της ζωής και αποφεύγουμε απώλεια ζώων. Και θεωρώ ότι αυτό ακριβώς το μήνυμά τους πρέπει να κατευθύνει ακριβώς το θέμα της δωρεάς των οργάνων, ώστε αυτά να, αυτή να προωθεί περισσότερο στις χώρες μέλη. Αλλά καταλαβαίνω ότι η Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες για να δράσει στον τομέα της δημόσιας υγείας. Και στις περισσότερες περιπτώσεις η δράση της Ένωσης περιορίζεται στην ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ τη δουλειά και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί, και να εφαρμοστεί η νομοθεσία που να θέτει υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τα ανθρώπινα όργανα. Οι διαφορές μεταξύ των χώρων μελών είναι πολύ σημαντικές. Υπάρχουν χώρες που εξαρτώνται πλήρω από διμερείς συμφωνίες, η χώρα μου είναι μία από αυτές και εδώ αναφέρομαι στη Μάλτα βέβαια, αλλά νομίζω ότι εδώ το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες μέλη, αλλά το θέμα της προώθησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχοντας κατά νου τις αρμοδιότητες της Ένωσης για αυτό το θέμα, να θυμόμαστε παρόλα αυτά και τις διαφορές μεταξύ των χωρών όπως μας είπαν στην παρουσίαση. Και το γεγονός ότι χρειαζόμαστε επίσης και μια αλλαγή στην δημόσια έτσι, στάση, στην στάση του κοινού, ώστε να έχουμε ακριβώς δηλαδή αύξηση σημαντική στην δωρεά των οργάνων αλλά και για τις ε, ζώντε δωρεές. Ε, για αυτό το θέμα θα ήθελα να καταλάβω περισσότερα από την Κομισιόν και να λάβω περισσότερες πληροφορίες. Καταρχάς για τις διασυνορικές συναλλαγές και κατά πόσο θεωρεί η Κομισιόν ότι αυτό πρέπει να βελτιωθεί και επίσης από τις κοπιές Κομισιόν να ακούσω ποια είναι η κυριότερη δράση που η Ένωση σφαιρικά και οι χώρε με μπορούν να αναλάβουν ώστε αν μην φτάσουμε στο μηδέν, τουλάχιστον να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται εν αναμονή, ώστε να μην έχουμε απώλεια ζωών μεταξύ των ατόμων που αναμένουν δηλαδή την τωρία οργάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Ανταλή. Ο κύριο Σελβενή, ο μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι καλή ευκαιρία νομίζω να συνοψίσουμε τη γνώση που υπάρχει γύρω, αυτό, από αυτό το θέμα. Και καταρχάς, εξωμάτως της ομάδας μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η οδηγία είναι χρήσιμη για να ενισχύσουμε την διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσουμε υψηλέ προγραφές ποιότητας όσον αφορά δωρεάν ανθρωπίνων οργάνων για μεταμόσχευση. Πέρασαν πέντε χρόνια από τη μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες και έχει σημειωθεί η πρόοδος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ζώσα δωρεά αποτελεί, συνεχίζει να αποτελεί μια συμπληρωματική πηγή που βασίζεται σε εθελοντική βάση. Και ε, ξέρω ότι ως θέμα είναι περίπλοκο. Αυτό το θέμα πρέπει βεβαίω να μας κάνει να σκεφτούμε για το θέμα της εμπορίας οργάνων. Της παράνομης εμπορίας οργάνων που δεν αποτελεί πρόβλημα εντό τη Ένωση, αλλά ξέρουμε ότι στην περιφέρεια της Ένωση είναι ένα απάνθρωπο εμπόριο και ανθυρό κιόλα και θα πρέπει να το προσέξουμε. Για την καταπολέμηση λοιπόν αυτού του φαινομένου αφαίρεση οργάνων και εμπορία τους, που είναι σημαντικό, θα πρέπει να πούμε ότι η χνηλασιμότητα αποτελεί το σημαντικότερο σημείο μαζί με την ασφάλεια βεβαίω για τους ενδιαφερόμενους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και στοχευμένο. Υπάρχουν και τα ατυχήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια των χειρουργείων και ξέρουμε τη σημασία τους και νομίζω θα υπογραμμίσω εν τέλει τη σημασία της εκπαίδευσης του εξειδικευμένου προσωπικού που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα δωρεάς οργανών. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εκπαίδευση όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, ώστε να στοχεύει στο συντονισμό της δωρεάς, κάτι το οποίο είναι μεγάλη σημασία. Αυτά τώρα για το γενικό κομμάτι και θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω κάποια πιο επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη χώρα μου. Και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Νομίζω ότι η οδηγία και η εφαρμογή της για τους ξένους δότες ή την έλλειψή τους, μας οδηγεί στο ερώτημα πώς εγκρίνεται η δωρεάν αυτή από ένα ξένο δωρητή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γραμμές στην Ένωση. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να ελέξουμε κατά πόσο ένας πολίτης ο οποίος είναι κλινικά νεκρός σε μια χώρα θα μπορούσε να δώσει όργανα ή όχι. Γιατί για το γεωγραφικό πεδίο δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εδώ περιθώριο ή ευχαίρια κινήσεων όσον αφορά αυτό το άτομο. Πρέπει να δούμε ακριβώς λοιπόν τι γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό, το, ατομικό επίπεδο και όχι σε γεωγραφικό. Και πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση επιτρέπουμε ή απορρίπτουμε την δωρεά και κατά πόσο αυτή τι απόφαση θα πρέπει να συνοδεύεται με το απαραίτητο έλεγχο βέβαια και την τεκμηρίωση. Αν λοιπόν μετά το θάνατο ενό ξένου επικόου υπάρχει ένα θέμα, πιθανό θέμα δωρεά, τότε η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της χώρας αυτού του επικόου και να εφαρμόσει βεβαίω τι ε, απαραίτητε νομικέ προδιαγραφέ εκείνη τη χώρα, ώστε να εγκριθεί τέλο πάντων η δωρεά αυτή. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο απόφασης θα μας επιτρέψει ακριβώς να έχουμε μια εποπτεία όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Ίσως να το θεωρείτε ακραίο σαν παράδειγμα, αλλά υπάρχουν πολλές χιλιάδες τέτοιων περιπτώσεων που κάθε χρόνο βλέπουμε να ανακέπτουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Ντορνάνο τώρα. dépit de l'intervention de l'Union από τη στιγμή που παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα όργανα που πάνε σε μεταμοσχεύσεις, να σας πω πως τα περισσότερα κράτη-μέλη απέκτησαν ε, συστήματα ε, που έχουν είτε ρητή, είτε έμεση, είτε υπονοούμενη ε, έγκριση. Και ξέρω πως το 20% μόνο των όσων έχουν ερωτηθεί είναι αρνητικοί στο να γίνουν δότες οργάνων, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κάπου να θεωρηθούμε ότι υπάρχει ε, σιωπηρή συγκατάθεση στην περίπτωση που δεν υπάρχει ε, πεφρασμένη αντίρρηση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αυξήσουμε ε, τις μεταμοσχεύσεις και να αποφύγουμε αυτή την, ε, το εμπόριο που γίνεται οργάνωση στην Ευρώπη που βασίζεται στην ε, οικονομική ανάγκη και στις χερίς συνθήκες που σε κάποιες κοινωνίες επικρατούν. Θα ήθελα τώρα το λόγο να δώσω στο λόγο και πάλι στον κύριο Σνίκελς για να απαντήσει στα σχόλια των όσων πήραν το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις πολύ καλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις. Κυρία Μάσινερ, ρωτήσατε για το εάν κάποιες χώρες, ε, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, ε, θα λάβουν μέρος. Η απάντηση είναι ότι όλες οι χώρες ε, συμμετέχουν στις συναντήσεις αρμοδίων αρχών και ομάδων εργασίας. Και όλες οι χώρες μπορούν να συμμετάσχουν και de facto το κάνουν. Παραδείγματο χάρη η Γερμανία ηγείται σε ένα από τα έργα που χρηματοδοτούνται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε έχει έναν πολύ ένεργο ρόλο στη, στα έργα αυτά. Τώρα γιατί υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Κύπρου, μάλλον για ιστορικούς λόγους, αλλά έχετε δίκιο, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην συνεργασία, το... ο χρόνος ε, ε, ζωής καρδιάς είναι 4-5 ώρες, ενώ ε, είναι πολύ μεγαλύτερος 24 ώρες ο χρόνος στον, κατά τον οποίο επιζεί ένα νεφρό. Αλλά αν δείτε την απόσταση μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου γίνεται. Και και βεβαίω μεταξύ Ιταλία και Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα και για καρδιές και πνεύμονες που έχουν σχετικά μικρή περίοδο επιβίωσης θα έλεγα. Μετά, ρωτήσατε για το σύστημα της συνένεσης. Ε, το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα ζητήματα ε, δεοντολογίας είναι εθνική αρμοδιότητα, οπότε είναι θέμα και πολιτισμού και κοινωνίας και αξιών να αποφασίσει κάθε χώρα και γεγονός είναι ότι έχουμε διαφορετικά συστήματα, έχουμε 17 χώρες με ένα σύστημα opt-out όπου πρέπει κάποιος να δηλώσει ότι δεν θέλει. Στη Γερμανία πρέπει να δηλώσει ότι θέλει και 4 χώρες με ένα μεικτό σύστημα. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν έχουμε διαφορετικά συστήματα τελικά στην πράξη οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, γιατί ακόμα και σε χώρες όπου προϋποτίθεται η συνένεση, κατά κανόνα έρχονται σε επαφή με τις οικογένειες. Και είναι νομίζω πολύ χρήσιμο αυτό, δηλαδή να δούμε το τι ε, είχε πει, τι επιθυμίες είχε εκφράσει ο δυνητικός δωρητής. Νομίζω πως είναι μια καλή αρχή αυτή που τηρείται παντού και αυτό κατά την απόψή μου εμέσως απαντά και στην ερώτησή σας γιατί κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, παρά το ότι είναι εθνική αρμοδιότητα να έρθουμε σε επαφή με την οικογένεια στην χώρα προέλευσης ή οπουδήποτε αλλού όπου η σύζυγος ή ε, ο σύζυγος ερωτούνται αν συμφωνούν με την δωρεά μετά. Υπήρχαν ερωτήσεις από την κυρία Νταλή και θα υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι στις λίστες αναμονής μεταξύ 50 και 60 και ακόμη χειρότερο πολλοί κόσμος πεθαίνει στη λίστα αναμονής ε, κατά μέσο όρο 4.000 ασθενείς ε, το έτος, κάτι το οποίο είναι πολύ προβληματικό. Το θέμα της λίστας αναμονής όμως το είχαμε συζητήσει και στην τελευταία συνεδρίαση. Είναι δύσκολο γιατί σε χώρες όπου έχουμε πολλές δωρεές οι γιατροί ε, είναι πιθανότερο να βάλουν τους ασθενείς σε λίστα αναμονής ενός χώρες όπου έχουμε δει μέσω σκανδάλων μία μείωση το ε, στο δωρητών, όπως στη Γερμανία, οι γιατροί δυσκολότερα θα βάλουν κόσμο στη λίστα αναμονής. Οπότε πρόκειται απλά για μια ένδειξη χωρίς ε, να λέει τα πάντα. Αλλά το ότι ο κόσμος πεθαίνει ενώ περιμένει στη λίστα αναμονής είναι προβληματικό και πρέπει νομίζω να μας ενθαρρύνει για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η στήριξή σας ως βουλευτές είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μιλάτε και με τους ε, δικούς σας τους ε, ψηφοφόρους ε, και ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Κοινοβούλιο είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα στις προσπάθειες στα κράτη-μέλη και οργανώνουμε εργαστήρια με δημοσιογράφους και καλό θα ήταν νομίζω και εσείς να πάτε σε αυτά τα εργαστήρια, να προωθήσετε την δωρεά οργάνων. Για τις διασυνοριακές ανταλλαγές έχουμε δύο ήδη, ε, πολυμερείς και διμερείς συμβάσεις. Στις πολυμερείς έχουμε τρία συστήματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Euro Transplant, Benelux, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Κροατία. Ε, το σκανδιναβικό σύστημα που είναι σκανδαλικές χώρες και η συμμαχία του Νότου, η Ιταλία, Γαλλία και η Ισπανία. Έχουν λοιπόν ανταλλαγές ε, οργάνων συστηματικές ε, με πολυμερείς ε, συμφωνίες που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Και από την άλλη έχουμε και διμερείς συμβάσεις και έχουμε αναπτύξει και ένα υπόδειγμα σύμβασης για να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των χωρών και αυτό νομίζω είναι ε, πολύ θετικό και βλέπουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτές οι συμβάσεις. Δυστυχώς δεν έχω τώρα πρόχειρα τα νούμερα, αλλά σε συστήματα όπως το Eurotransplant και το Scania Transplant βλέπουμε συστηματικά να πηγαίνουν τα όργανα από το Βέλγιο στη Γερμανία ή στην Αυστρία και αντιστροφώς. Μετά είχαμε ένα ερώτημα το οποίο αφορά τις εθελοντικές δωρεές και την παράνομη διακίνηση. Εμείς έχουμε συμφωνήσει με τις εθελοντικές δωρεές χωρίς πληρωμή που είναι το αντίθετο από την παράνομη διακίνηση. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη και αν δείτε το ζήτημα πιο στενά θα δείτε ότι υπάρχουν ασθενείς που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν μία μεταμόσχευση και μετά επιστρέφουν ε, και βλέπουμε επίσης ότι οι ασθενείς αναζητούν όργανα στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά μέσα και κάνουν ακόμα και προσφορές. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι περίπλοκη, αλλά το καλό είναι ότι όλες οι αρμόδιες αρχές ε, επαγρυπνούν και μόλις έχουν μία ένδειξη κινητοποιούνται. Και αυτό είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε ε, πέρα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση. Θετικό επίσης είναι ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εγκρίνει μία συμφωνία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προετοιμάζει μία σχετική δήλωση έτσι ώστε υπάρχει η αρχή παγκοσμίω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πληρωμή για δωρεά οργάνων. να, πρέπει να επαναλάβω αυτό το οποίο είπατε για την κατάρτιση. Έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει κάποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συντονιστές μεταμόσχευσης είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο με την Ολλανδία και την Ουγγαρία, όπου οι χειρουργοί εκπαιδεύτηκαν από πολύ έμπειρους Ολλανδούς ε, χειρουργούς και δημιούργησαν ένα βίντεο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ε, χώρες ε, για το πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα αυτές οι δωρεές οργάνων. Μετά υπήρχε ένα ερώτημα από τον κύριο για τα συστήματα συνένεσης και το ότι 80% των πολιτών συμφωνούν πράγματι, ισχύει αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επισημάνω το ότι βεβαίως ε, το ποσοστό δωρεών εξαρτάται όχι μόνο από την συνένεση αλλά και από ολόκληρο το σύστημα που υπάρχει. Να σας δώσω το παράδειγμα της Γερμανίας όπου επίσης έχουμε πολύ υψηλή συνένεση του 80% των ανθρώπων. Παρόλα αυτά είδαμε δραματική πτώση στις δωρεές γιατί λόγω των σκανδάλων και ο κόσμος ε, στα νοσοκομεία πλέον δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή λένε όταν ε, ε, ξεκινήσω με τέτοιο, κινδυνεύω να μπλέξω σε ένα σκάνδαλο. Οπότε δεν λέω καν ότι έχω ένα ασθενή που είναι δυνητικό δωρητή. Οπότε είναι σημαντική συνέντευξη, αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να υπάρχει. Οπότε το σύστημα της συνένεσης δεν είναι τόσο αποφασιστικό για το ποσοστό δωρεών. Για τα ζητήματα παράνομης διακίνησης ε, τα απάντησα ήδη, νομίζω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που προτείνω τώρα είναι, εάν δεν ζητάει κανείς το λόγο, να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Είναι το σημείο 5 της ημερής διάταξης που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων παρακολούθησης των κρατών μελών βάσει της οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο κύριος Φρανσουά Βάκενχουτ, διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον, στη Διεύθυνση ε, ΓΑΜΑ ποιότητα ζωής. Έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι πραγματική χαρά που έχω τη δυνατότητα να λάβω το χώρο, το λόγο με συγχωρείτε εδώ, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που έχουμε ε, για την παρακολούθηση των κρατών μελών βάσει της οδηγίας πλαίσια για τη θαλάσσια στρατηγική και βάσει ε, της ε, στρατηγικής που ε, ενέκρινε και υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιανουαρίου τρέχοντος. Θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία η οποία προβλέπεται στα πλαίσια της, του, της οδηγίας σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν θαλάσσιες στρατηγικές. Αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ε, νομοθεσίας μας και βεβαίως αυτές οι στρατηγικές αξιολογούνται κάθε έξι χρόνια. Θα δείτε την διαφάνεια που αναφέρεται στα βήματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια τέτοια θαλάσσια στρατηγική. Καταρχήν, μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη ε, και πώς έχουν οι θάλασσες εκεί. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Μετά, ορίζεται αυτό που εμείς ε, ονομάζουμε στην οδηγία η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως επίσης και οι στόχοι. Δηλαδή τι προσπαθούμε να πετύχουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτά τα θαλάσσια συστήματα, τα οποία εξαρτώνται από το θαλάσσιο περιβάλλον. Μετά έχουμε τα προγράμματα παρακολούθησης και τέλος χρειάζεται να εντοπίσουμε και να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο δράσεων που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε αυτή την καλή περιβαλλοντολογική κατάσταση, το GIS. GES, με Θα παρουσιάσω τους στόχους από σήμερα το απόγευμα και στη συζήτηση που θα κάνουμε θα σας πω τι έχουμε εξετάσει εμείς ε, σε επίπεδο προγραμμάτων κρατών μελών. Καταρχής, κατά πόσο είναι ενδεδειγμένα, είναι κατάλληλα για να ελέγξουν τον την πρόοδο που έχουν κάνει στο θαλάσσιο περιβάλλον έτσι ώστε να πετύχουν τον στόχο του καλού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην αξιολόγηση που κάναμε διαπιστώσαμε πως έχουν κάνει πολλές προσπάθειες στα κράτη-μέλη, κάτι το πολύ θετικό, Όμω η έκθεση αποδεικνύει πω χρειάζεται περαιτέρω δράση στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως έχουμε την κατάλληλη και την έγκαιρη παρακολούθηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Το συμπέρασμα είναι πως κανένα από τα προγράμματα είναι απολύτως, δεν είναι απολύτως κατάλληλο για να πετύχει τους στόχους της οδηγίας, δηλαδή παρακολούθηση της διαδικασίας και των στόχων έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτό το καλό περιβάλλον. Και στην διαφάνεια εδώ σας δείχνω πως η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Λετωνία έχουν προγράμματα παρακολούθησης τα οποία δεν είναι κατάλληλα πάντα αξιολογημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε. Η Βουλγαρία, κάτω χώρες, Ισπανία και η Φιλανδία έχουν αναπτύξει προγράμματα που είναι κατά μεγάλο ποσοστό ενδεδειγμένα, δηλαδή εδώ εξετάζουμε αυτούς που αποδίδουν περισσότερο και όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα υπόλοιπα προγράμματα παρακολούθησης είναι στη μεσαία κατηγορία των μερικώς ενδεδειγμένων προγραμμάτων. Βλέπετε λοιπόν και εσείς πως αυτό που έχουμε πετύχει είναι μία μάλλον μεικτή απόδοση και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σίγουρα χρήζει βελτίωσης. Να περάσω λοιπόν στο επόμενο που είναι ένα επίσης σημαντικό συμπέρασμα από την έκθεση που είναι πως τα προγράμματα παρακολούθησης των κρατών μελών δεν ήταν άμεσα λειτουργικά. Το 2014 μόνο μερικοί τα είχαν ήδη στήσει και κάποια θα είναι στη θέση τους μόνο το 2018 και κάποιοι θα πάνε και στο 2020 για να ετοιμαστούν. Αυτό βεβαίως προκαλεί προβλήματα γιατί κατόπιν πρέπει να μετρηθεί και η πρόοδος όπως επίσης και η απόδοση και οι επιδόσεις. Επίσης, το πεδίο της παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση είδε πως παρακολούθηση κάποιων στοιχείων που είναι πολύ συγκεκριμένα για την οδηγία μας όχι μόνο παρακολουθούνται από άλλη νομοθεσία, αλλά παρακολουθούνται με έναν τρόπο που δεν είναι κατάλληλο και θα σα δώσω παραδείγματα. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, ο υποθαλάσσιο θόρυβο, ε, τα μη η, τα γεννή φυτά, όπω επίση τα θαλάσσια απορρίμματα. of the marine environment are directly linked και τις άλλες πτυχές του θαλασσίου περιβάλλοντος που σχετίζονται άμεσα με την άμεση εφαρμογή άλλης νομοθεσίας, όπως παραδείγματο χάρη τον κανονισμό για τα αυτόχθονα είδη. Λοιπόν, πού πάμε ε, από εδώ και προς. Με βάση την ανάλυση που έχουμε κάνει, η Κομισιόν επίσης προσπαθεί να κάνει κάποιες γενικές συστάσεις και κάποια κατεύθυνση προς τα κράτη-μέλη για να εστιάσουμε ότι θα υπάρχει η σωστή παρακολούθηση και θα καλύπτει όλα τα, όλες τις περιγραφικές πτυχές ε, και τις επιχειρησιακές, το συντομότερο δυνατόν. Έτσι καταλήξαμε στο ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τα εξής. Πρώτα απ' όλα να δούμε το συντομότερο δυνατόν τις ελλείψεις που έχουμε δει σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε τα προγράμματα παρακολούθησης είναι τα κατάλληλα για να επιτευχθούν οι απαιτήσει που ορίζει η οδηγία πλαίσιο. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εφαρμόσουν πλήρως τα προγράμματα παρακολούθησης για να και να στην ε, αξιολόγηση των θαλασσιών υδάτων το 2018, του χρόνου δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση της απόφασης 2010 για 2010 καθώς 44 καθώς 7 καθώς Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτύχουν μεγαλύτερη συνοχή στο περιφερειακό ή επίπεδο μέσω περαιτέρω συντονισμού των προγραμματών παρακολούθησης κυρίως μέσω κάποιων βασικών στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή της ε, οδηγίας, ε, την συνεργασία με τη Συμβάση για την Θάλασσα και βεβαίως ε, κοινέ προσεγγίσεις για συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων. Η Κομισιόν λοιπόν σκοπεύει να κάνει περισσότερα η ίδια για να επιταχυνθεί ο ρυθμός εφαρμογής και να έχουμε αποτελέσματα συγκεκριμένα. Η Κομισιόν θα στηρίξει τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα αναζητώντας συνέπεια στην εφαρμογή ε, διαφόρων ε, τμήματων της κοινωτικής νομοθεσίας που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό θα γίνει κυρίως αναθεωρώντας την άποψη που ορίζει τα κριτήρια και την μεθοδολογία για, το, ε, καλό, για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, κάτι το οποίο θα γίνει σύντομα από την Κομισιόν. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε την συνεργασία με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο μιας εντατικής διαδικασίας, ε, στο πλαίσιο της κοινή στρατηγικής εφαρμογής ε, της οδηγίας πλαισίου, που είναι το γενικότερο πλαίσιο για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Τρίτον, θα εξετάσουμε την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης στρατηγικών έργων ε, και δράσεων υποστήριξη για να διευκολύνουμε την συνέπεια στο επίπεδο περιφερειών και ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσια. Επίσης θα οργανώσουμε διμερείς συναντήσεις με τα κράτη-μέλη εκείνα, τα προγράμματα των οποίων θεωρούνται μη κατάλληλα και βεβαίως ε, θα συνεχίσουμε την ε, παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται στα κράτη-μέλη. Το επόμενο βήμα μετά τα προγράμματα παρακολούθησης είναι τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αναφορές προς την Κομισιόν τα προγράμματα μέτρων που έχουν σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως μόνο 16 κράτη-μέλη έχουν αυτή τη στιγμή ενημερώσει την Κομισιόν σχετικά. Περιτώ να πω ότι άρα ε, έχουμε πει στα κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα να μας κοινοποιήσουν το συντομότερο δυνατό τα αποτελέσματα. Ε, Προσπάθησα να είμαι σύντομο κύριε Πρόεδρε, δεδομένου του χρόνου που έχουμε. Ε, ελπίζω λοιπόν η παρουσίαση που έκανα να σας έδωσε μία εικόνα των εξελίξεων μέχρι στιγμής για τα προγράμματα παρακολούθησης και για τις γενικές κατευθύνσεις για το βασικό νομοθετικό όργανο που έχει αναπτύξει η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους οι οποίοι μας ζήτησαν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Νταλή πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και για μια φορά ακόμα θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πραγματικά ε, αυτό το θέμα το έθεσε στην κορυφή της ε, ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ είμαι από, από ένα μικρό νησί στη μέση τη Μεσογείου, οπότε το γεγονό ότι συζητάμε το θέμα αυτό ε, έχει να κάνει με συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο στη χώρα μου. Θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για τα θαλάσσια απόβλητα, θαλάσσια απορρίμματα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ε, επί των οποίων χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Το θέμα που προκύπτει και νομίζω ότι εδώ θα ήθελα να εστιάσω είναι το γεγονός πως, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανένα από τα προγράμματα παρακολούθησης δεν είναι απολύτως ενδεδειγμένο και κάποια είναι μόνο εν μέρη ενδεδειγμένα. Όταν εγώ διάβασα την έκθεση, μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο σημείο που με ενδιέφερε είναι το γεγονός πως αρκετά σημεία χρειάζονται ε, αμέσως βελτίωση και πιο συγκεκριμένα τα θαλάσσια και ο τρόπος με τα οποία τα παρακολουθούμε, τι γίνεται με τα απόβλητα στο βυθό και η παρακολούθηση των μικροαποβλήτων ή μικροαπορριμμάτων, όπου και εκεί δεν είναι κατάλληλη η παρακολούθηση. Με ανησυχία διάβασα πως δεν υπάρχει συστηματική και συγκριτική ανάλυση του πώς επηρεάζουν αυτά τα απορρίμματα τους ανθρώπους και τα ζώα. Όπως επίσης το τι συμβαίνει ε, με τα απόβλητα που δημιουργεί ο άνθρωπος ε, και που καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας. Επίσης, είπατε μερικώς ενδεδειγμένα. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγκεκριμένα ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτή τη μερική εφαρμογή Ξέρω πως αναφερθήκατε σε κάποιους κλάδους όπου υπάρχουν άμεσες συνέπειες, αλλά ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραπάνω στοιχεία. Επίσης, οι συστάσεις που θα υποβάλλετε, κατανοώ την εξήγηση που δίνετε για το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παρακολούθηση ε, ε, τα κράτη-μέλη με περιφερειακά ή διαπεριφερειακά προγράμματα. Αλλά αυτές οι γενικές συστάσεις πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη είναι αρκετά δύσκολο για κάποια κράτη-μέλη. Και αν ισχύει αυτό, μήπως επιβαρύνουμε κάποια κράτη-μέλη υπερβολικά. Το ρωτώ γιατί θέλω να καταλάβω καλύτερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όπου θα έχουμε προγράμματα παρακολούθηση τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα. Και επίσης μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως μόνο 16 κράτη-μέλη υπέβαλαν τα προγραμματά τους μέχρι σήμερα. Ξέρω, όπως είπατε κι εσείς, πως είστε σε επαφή με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αλλά πείτε μου, τι θα συμβεί. Έχετε προβλέψει κάποιες ε, καταληκτικές ε, προθεσμίες, προσπαθείτε να εξασφαλίσετε πως θα τα λάβετε μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποια είναι τα επόμενα σας βήματα. Επίσης, τέλος, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική κατά τη γνώμη σας για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το κίνδυνο για την, δημόσια, την ανθρώπινη υγεία, για την υγεία των θαλασσίων οργανισμών, όπως επίσης για τα μικροαπορρίμματα και για τα θαλάσσια απόλυτα και απορρίμματα που καταλήγουν στο βυθό. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος uh, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Έχω την εντύπωση ότι συχνά κάποιες ε, νομοθετικές προτάσεις υπογράφονται από τα κράτη-μέλη και μετά δεν τηρούνται. Αυτό είναι το πρόβλημα και εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, τα θαλάσσια και εκεί πέρα συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα, αυτό το πράγμα και είναι λυπηρό γιατί ακριβώς έχει μεγάλη σημασία για να είναι καθαρές ή να ξαναγίνουν καθαρές οι θάλασσες και να εμποδίσουμε τα χειρότερα στο μέλλον. Γι' αυτό έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το πρώτο, πολύ καλή η παρουσίασή σας, μπορείτε να μας την ε, στείλετε. Καλό είναι να την έχουμε. Το δεύτερο ερώτημα, μέχρι πότε πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία, δεν το είπατε. Ε, και θα θέλαμε να δούμε, υποθέτω ότι έχει περάσει και θα έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί. Τρίτη ερώτηση για την παρακολούθηση. Είπατε ότι υπάρχουν λίγες χώρες που τα εφαρμόζουν λογικά. Και βεβαίως έχουμε και την ε, Πορτογαλία η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα αλλά στην οδηγία δεν ε, οριζόταν τι μορφή θα έχει η παρακολούθηση. Δηλαδή, κατά κανόνα υπάρχουν οι πράξεις κατευσιοδότηση ή άλλες διατάξεις ε, για να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Μετά το επόμενο ερώτημα με τα κράτη-μέλη. Η κυρία Ντελή είπε τι κάνουμε για να το ακολουθήσουν και άλλοι. Ε, μπορούμε να έχουμε τον κατάλογο. Γιατί θα ήθελα να δω ποια κράτη-μέλη το έχουν εφαρμόσει και ποια όχι για να μπορέσουμε και εμείς να ασκήσουμε κάποια πίεση στα κράτη-μέλη που δεν αντιδρούν. Και τελευταία ερώτηση. Ε, για την ε, περιφερειακή συνεργασία έχουμε ε, αποφασίσει τόσο πολλά προγράμματα για το θαλάσσιο περιβάλλον ε, ώστε θα έπρεπε να λειτουργεί κάτι τέτοιο. Μήπως λοιπόν τα κράτη-μέλη γενικώ δεν θέλουν να μπλέκεται πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα των ακτών, γιατί είχαμε και τον κανονισμό της ε, θαλάσσιας χορταξίας, δεν ήθελαν καθόλου την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών ε, και είχα την αίσθηση ότι και το MSFD πραγματικά ε, τους ήταν αδιάφορο. Κάνω λάθος ή όχι. Σας ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Δίνω τον λόγο τάσο, κύριο Φόντε. Ευχαριστώ. Η έκθεση αλλά και η παρουσίαση, έστω και συντομότερη, προσιάζει μια εικόνα ανησυχητική. Είδαμε επανειλημμένως να έχουμε καλή στρατηγική και οδηγία και φιλόδοξη, αλλά μετά το μπαλάκι πάει χώρε μέλη και αρχίζουν τα προβλήματα. Τότε με αυτό με την στρατηγική για την βιοπικιλότητα, όπου η μεσοπρόθεσμη στρατηγική ήταν καταστροφική και το ίδιο βλέπουμε επίσης για αυτή την θαλάσσια στρατηγική, όπου έπρεπε να περιοριστούμε, περιοριστούμε τρόπος του λέγει μόνο στην παρακολούθηση και στην εποπτεία. Έχουμε τις προθεσμίες του 18 και του 20 που πλησιάζουν και η εικόνα πραγματικά είναι απογοητευτική για την οδηγία. Να τονίσω δύο ζητήματα συγκεκριμένα τώρα. Πρώτον, όσες χώρες έκαναν κάτι, το έκαναν. Άλλες ήταν πιο αργές και χρησιμοποίησαν διατάξεις και τρέχουσες δράσεις τις οποίες συνέχισαν αλλά εκεί που χρειαζόταν νέες δράσεις νέες ιδέες μεγαλύτερη προσπάθεια κτλ. για να υλοποιηθούν καινοτόμα προγράμματα, αυτό δεν έγινε, δεν υπήρξε. Και αυτά τα δύο θέματα που αποτελούσαν τη βάση τη θαλάσσιας στρατηγική δεν υλοποιήθηκαν στην ουσία καθόλου. Οι προτάσει τώρα της Κομισιόν για παρεμβάσεις, εντάξει σημαντικέ είναι, αλλά νομίζω ότι δεν επαρκούν και χρειάζεται όθηση και δέσμευση μεγαλύτερη. Και κάτι άλλο που ανέφερε σαν αφός Ντάλι και το ξαναλέω, τα απορρίμματα, τα θαλάσσια, που πρέπει στο πλαίσιο της ανακοίνησης Κομισιόν να δοθεί ιδιαίτερη έφαση, αλλά ξαναλέω, για την επιφάνεια, για το βυθό κτλ. Έχουμε στοιχεία, αλλά μας λείπουν στοιχεία, ας πούμε, για την ε, θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Βέβαια, αυτό βρίσκουμε και στο Ocean Governance, στην θαλασσία διακυβέρνηση, η διακυβέρνηση των, ωκεα... των στην ε, γαλάζια οικονομία. Και βλέπουμε ότι και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των λιγιών για την κυκλική οικονομία. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει δραματικό με πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Επιπτώσεις τις οποίες κάποιες από αυτές μόλις τώρα συνειδητοποιούμε. Ίσως λοιπόν εδώ η Κομισιόν έπρεπε να τολμήσει περισσότερο να συνεχίζει να πιέζει τι χώρε μέλη βέβαια, αλλά διαρωτώ με μήπω θα έπρεπε πραγματικά να γίνει μια πραγματική παρέμβαση για τα θαλάσσια αυτά ζητήματα, ισχυρή παρέμβαση, νομοθετική. Και τέλος, να ρωτήσω το εξή. Στο Ocean Governance μιλάμε για τα θαλάσσια παρέμβατα, για να θεώρηση των κανονισμών των λιμένων, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της αλίας για την ανάκτηση αυτών των απορριμμάτων. Θα ήθελα να μου το βεβαιώσετε αυτό γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος να το διευθυντής και πάλι. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις σημαντικές ερωτήσεις μετά την έκθεση και την παρουσίασή μου. Να ξεκινήσω για το πρώτο, τα θαλάσσια απορρίμματα που αναφέρθηκαν επαγγελμένως και θα αναφέρω σε αυτό εκτενώς. Τώρα για τις γενικές συστάσεις και το αντικτυπώ τους και το follow-up είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε ενεργά. Και πολύ ενεργά θα παρακολουθήσουμε με τις χώρες μέλη την εξέλιξη των προγραμμάτων τους. Θα έχουμε διμερείς συναντήσεις με αυτές τις χώρες τους ερχόμενους μήνες για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες να βελτιώσουν τα προγράμματά τους εν ώψη του νέου κύκλου που θα ξεκινήσει το 2018 και επίσης ενεργά θα κινητοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε υπό την κοινή στρατηγική. Αυτά για να σας αποδείξω το ότι πραγματικά κάναμε παρατηρήσεις στην έκθεση και προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε. Και αυτό είχε σχέση με αυτό που είπατε την πρόοδο στι διάφορε χώρε μέλη, ίσω βουλευτέ. Τώρα για τα προγράμματα με μέτρα και το γεγονό ότι 16 χώρε μέλη υπέβαλαν εκθέσει για τα προγράμματά του. Να σα πω ότι έχουμε ξεκινήσει διαδικασίε παραβίαση. Έχουμε ξεκινήσει για όσα εξέπνευσαν 31 Μαρτίου 2016. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίε παραβίαση ε, το Φεβρουάριο του 2017 φέτος δηλαδή, το οποίο αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν σε περιπτώσει όπου τα πράγματα δεν πάνε ικανοποιητικά. Να πω κάτι και για το χρονισμό της εφαρμογής, για το οποίο είχαμε δύο ερωτήσει. Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 20, ως ονούπο δηλαδή. Αν δείτε και την έκθεση πρόοδου, αυτό είναι προφανές ότι θα πρέπει τα πράγματα να επιταχυνθούν αν θέλουμε να το πετύχουμε. Και η Κομισιόν θέλει να γίνουν όλες οι απαραίτητε προσπάθειες ώστε να τηρήσουν την προθεσμία 2020. Τώρα, για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην, στην Πορτογαλία, είχα μια επί τούτου ερώτηση. Οι ΑΟΣ και οι θαλάσσιες περιοχές της ε, Πορτο... Πορτογαλίας παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Πάντως, είδαμε ότι το επίπεδο συμμετοχής και οι δράσει δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Ίσως να υπάρχει ένα θέμα μεγέθους προσπάθειας. Περιφερειακή συνεργασία. Αυτό υπάρχει και εφαρμόζεται. Οι συμβάσει περιφερειακών θαλάσσων, με περιφερειακή συμβάση για τη θάλασσα, μας παρέχουν το πλαίσιο ακριβώς για να εντατικοποιήσουμε τις προσπαθίες μας. Ε, και θεωρώ ότι είναι νωρί για να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε βέβαια την ενεργό συνεργασία υπό τι συνθήκε αυτέ, ώστε να πετύχουμε τα σωστά αποτελέσματα για τις περιφερειακές μας θάλασσε. Και σε αυτό ακριβώ δουλεύουμε, ώστε να υπάρχει συνέπεια με το σχεδιασμό που αναφέρατε και εσεί προηγουμένω και το εργαλείο που έχει αναπτυχθεί γι' αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό βέβαια. Τώρα, για τις ανεπάρκειες των μέχρι τώρα προσπαθειών και τις παρενέργειες μέχρι το 20. Να σας πω ότι η ειδικοποίηση των προσπαθειών είναι απαραίτητη για να πετύχουμε το αποτέλεσμα τώρα για τα θαλάσσια απορρίμματα συγκεκριμένα που αναφέρθηκαν από διάφορους ομιλητές. Τι κάνουμε γι' αυτό το θέμα εμείς. Κάνουμε πολλά να σας πω. Και μέσω TMSFT, αλλά και μέσω του πακέτου νομοθεσίας, αλλά και ε, μέσω της νομοθεσίας που αφορά τα απορρίμματα στους λιμένες. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε μια στρατηγική για τα πλαστικά. Τμήμα του πακέτου της κυκλικής οικονομίας. Προσπαθώντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα μάκρο και τα μικρο απορρίμματα. Και τους ερχόμενους μήνες θα κάνουμε διάφορες δράσεις με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών γιατί δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα των απορριμμάτων, όχι μόνο στην Ένωση, αλλά και στην γειτονιά της και παγκοσμίω. Υπάρχουν πολλές δράσεις λοιπόν οι οποίες γίνονται, τουλάχιστον μέσω των συμβάσεων περιφερειακών θαλασσών, αλλά και σε επίπεδο G20 και σε επίπεδο βέβαια διακυβέρνησης των θαλασσών που αναφέρθηκε προηγουμένω. Τώρα για τις δράσεις συγκεκριμένα σε αυτό το πλαίσιο αυτή την νέα μας απόφαση, τα κριτήρια των χωρομελών θα πρέπει να θεσπίζονται πιο ακριβέστερα, με πιο ακριβή τρόπο. Αυτό δεν είναι αμεληταίο και θα σας εξηγήσω. Αυξάνονται και τα μικρο και τα απορρίμματα. Αυτά που είναι αντικείμενο κατάποση από διάφορα ζώα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και τις κατάλληλες μεθόδους παρακολούθησης και αυτό νομίζω αποδεικνύει και τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς, ακριβώς αναγνωρίζοντα τη σημασία που έχει αυτό το θέμα. Να τονίσω επίσης ότι ενώ δεν μπορούμε να υποτιμάμε το ότι τα απορρίμματα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το θαλάσσιο περιβάλλον, εμείς θα πρέπει να παραβλέπουμε τις πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες προέρχονται από την ανηλία και από τις ζημίες στο βυθό της θάλασσας. Κάτι το οποίο απαιτεί βεβαίω και σοβαρές προσπάθειες αν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Τώρα σχετικά με τη μείωση της βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον στην περίοδο εφαρμογής πρέπει να σας πω ότι η εποπτεία είναι κρίσιμη σημασία ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις αυτού του θέματος. Και εδώ ακριβώς θα κρυθεί και η αξιοπιστία μας όσον αφορά τα, τις επιδόσεις μας. Σε εσείς είναι καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν να λάβουμε την απαραίτητη γνώση η οποία θα μας βοηθήσει ακριβώς στην φάση της εφαρμογής. Αυτά είχα να σας πω εγώ κυρίως και είμαι στη διάθεση να απαντήσω οποιοδήποτε άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Διευθυντά για τις απαντήσεις αυτές που δώσατε. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε άλλους που ζητούν το λόγο, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6, που είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση ε, CE στην αγορά αυτή τη στιγμή λοιπόν θα, εξετάσουμε το κείμενο και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Γκαρντίνη που είναι η εισηγήτρια. Συντέντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω βαρχνιάσει να με συγχωρείτε. Εδώ και ένα δεκαήμερο μετά από αυτή τη ζεστή εβδομάδα που είχαμε και το air condition. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή των εργασιών. Έχουμε και συνάντηση των σκιωδών απόψε και ίσως μετά να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε περισσότερους συναδέλφους. Όπως ξέρετε συζητάμε αυτή την πρόταση κανονισμού που διευρύνει ακριβώς το πεδίο για αυτά τα προϊόντα με σήμα ένωσης για να αντικατασταθεί και ο τερνός κανονισμός που αφορά τα προϊόντα αυτά λίπανσης από πρώτες ύλες. Ελπίζω να εφαρμοστεί σύντομα ώστε να επιτρέψουμε την είσοδο στην αγορά όχι μόνο προϊόντων λίπας, αλλά και να ελοποιήσουμε την οικονομία την κυκλική και τις αρχές της. γιατί θεωρούμε ότι αυτό βεβαίω θα ενισχύσει και θα προωθήσει και τις επενδύσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ε, κυκλική οικονομίας. Θα σα κάνω τώρα μια επισκόπηση της κατάστασης. Βρισκόμαστε στην αρχή. Και είναι πυκνή η δουλειά μας στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, γιατί έχουν καταφτάσει πολλές τροπολογίες. 711, εκτός αυτές της εισηγήτριας, με προθεσμία 7 Μαρτίου. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά γιατί για το κάδμιο ας πούμε και τα όρια έχουμε πολλή δουλειά επειδή υπάρχουν θέσεις αποκλίνουσες και αντικρουόμενες οπότε οι σκιώδεις θα πρέπει να αναζητήσουν κάποιους συμβιβασμούς αν έχετε προτάσει από αυτό λοιπόν παρακαλώ να τις υποβάλλετε γιατί το θέμα είναι αρκετά λεπτό όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία, για το κάσμιο και τα ωριά του. Πάντως έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά μας πάνω σε 8 συμβαστικές προτάσεις που αφορούν κάποιες θεματικές. Τέσσερις από αυτές τις συμβαστικές προτάσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, απλά και μόνο αποτελούν ένα σχέδιο, ένα μάλλον προσχέδιο ανοιχτό σε αλλαγές και παρατηρήσεις. και ελπίζω τέλο πάντων να καταλήξουμε σε μια δουλειά χρήσιμη για όλους. Πάντως οι πρώτες τέσσερις, ξαναλέω, αφορούν τους δρύπους, τους μικροβιακούς διαφόρων κατηγοριών. σε σχέση με τα προϊόντα λίπανσης και τα οργανικά δηλαδή και τους τροποποιητές και τα προϊόντα εξαγωγής των ε, καλλιεργιών. Προσπάθησα πάντως με βάση το κείμενο της Κομισιόν να διευκρινίσω ακριβώς το όριο αυτών των παθογόνων παραπέμποντας βέβαια στο οργανισμο 142 142-2010 που αφορά βεβαίω τα προϊόντα ζωικής προέλευσης κάτι το οποίο βεβαίω είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί αφορά βεβαίως και τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Και αφορά επίσης κάποια δείγματα τα οποία δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα. Αυτό είναι λοιπόν το περιεχόμενο των τεσσάρων πρώτων ε, συμβαστικών προτάσεων πάνω στους οποίες δουλεύουμε. Μετά έχουμε άλλο ένα σχέδιο συμβασμού σε σχέση με την χρήση άλλων προϊόντα που είναι ανακτήσιμα, όπως προϊόντα με βάση στάχτης. Πάντως αυτό που θα θέλω να διευκρινίσω είναι ότι μεταξύ των απορριμμάτων τα οποία επανακτώνται και που αφορούν την 2008-98 οδηγία, αυτή που φορά δηλαδή τα απορρίμματα, μεταξύ αυτών λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων λίπανσης αυτά τα προϊόντα, όπως σας έλεγα, δύο-τριών κατηγοριών, μεταξύ άλλων και τα προϊόντα της στάχτης, που σε κάποιες χώρες μέλη δεν ε, αδειοδοτούνται ή δεν επιτρέπονται από εθνικές νομοθεσίες. Για να δώσουμε λοιπόν κίνητρο στα πλαίσια πάντα της κυκλικής ε, οικονομίας, ζητάμε ακριβώς και την διεύρυνση της λίστας ε, για να ενταχθούν ε, προϊόντα τα οποία αφορούν ε, ανάκτηση, αφορούν προϊόντα απορριμμάτων με σήμανση ΕΕ και τα οποία ανακτώνται. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μέσω κατοξιδότηση πράξεων της Κομισιόν που θα μπορούσαν να θεωτηθούν βεβαίως μετά από την θέση ισχύ του κανονισμού. Πάντως δεν χρειάζεται να παραλάβω εδώ ότι οι κατοξιδότηση πράξεις στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημαντικές ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο εμείς διασφαλίζουμε το ότι η τεχνολογική εξέλιξη εφαρμόζεται και ότι δεν υπάρχει ένα είδος έτσι, παράτασης ή καθυστέρησης με άλλες διαδικασίες, άλλες διαδικασίες εκτός δηλαδή της πράξεων, ώστε να επιτρέψουμε μια ταχεία και γρήγορη εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Μετά έχουμε επίσης για τα οργανικά προϊόντα εσείς Λέμε ας πούμε ότι ο άνθρακας θα πρέπει να είναι οργανικός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σχετίζεται ας πούμε με το ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του προϊόντος λίπανσης στην παραγωγικότητα του εδάφους. Και μετά αναφερόμαστε σε τρία συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία αυξάνουν ακριβώς την απόδοση του εδάφους. Χωρίς παρενέργειες στο περιβάλλον. Νομίζω θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, χρήση μη αποτελεσματικών λιπασμάτων. Και έχουμε επίσης να σας πω και μια περιγραφή των ε, οργανικών και ορυκτών λιπασμάτων, τα οποία αποτελούνται από πάνω από ένα συστατικά. Ε, η Κομισιόν είχε αναφέρει στην αρχή ένα μόνο συστατικό, αλλά μετά από διάφορες μελέτες που κάναμε, βλέπαμε ότι αυτό δεν ήταν τεκμηριωμένο περιβαλλοντικά για λόγους υγείας και η επιλογή μιας μοναδικής και μόνο ουσίας περιόριζε ακριβώς την γάμα προϊόντων ή ουσιών που ήταν διαθέσιμα ή διαθέσιμα στους γεωργούς. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό εδώ να περιλάβουμε τους ε, βιολογικούς παράγοντες όπως αυτούς που λέγαμε προηγουμένως των τριών κατηγοριών. Μετά έχουμε επίσης και τα φυτά τα οποία είναι αντικείμενο μηχανικής επεξεργασίας ή εχειλίσματα φυτών και προσπαθήσαμε εδώ ακριβώς να κάνουμε πιο διεξοδικό το κείμενο της Κομισιόν. Τα φυτικά χιλίσματα και τα προϊόντα διαδικασίας εκχυλίσματος επεκτείνονται σε τέτοιο σημείο ώστε το πλέον αυτό να μην υπόκειται στις υποχρεώσεις του κανονισμού REACH. Και ξαναλέω, μόνο οι πρώτες τέσσερις συμβαστικές ε, προτάσεις αφορούν όλα αυτά τα θέματα. Τα, υπόλοιπα τέσσερα συμβαστικά σημεία συμβασμού είναι σημεία τα οποία αφορούν το παράτημα 1 και 2 σε συνεργασία με άλλες επιτροπές, άγκρι κλπ και αφορούν βεβαίω τα σημεία κοινή αρμοδιότητα, τα οποία δεν θα σα αναφέρω βέβαια ε, τώρα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τι ε, ανταλλαγέ σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Τώρα για το τμήμα που είναι καθαρά αρμοδιότητα έμβη, η πρόκληση θα είναι βεβαίω να βρούμε ένα συμβασμό για τα όρια καδμίου για αυτά τα προϊόντα λίπανσης όπου η κατάσταση είναι κακή. Αλλά ξέρετε ποια είναι η θέση μου. Θέση η οποία ήταν ακριβώς για να ξεκινήσει ένας διάλογος, επειδή θεώρησα ότι ήταν σημαντικό στους συμβασμούς να λάβουμε υπόψη μας δύο θέματα τα οποία δεν αποτελούν ακόμα ισχυρές πεπιθήσεις. Γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας σε σχέση με το κάδμιο που βρισκόμαστε. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, όπως επίσης δεν έχουμε αντιμετωπίσει και την ε, διαχείριση του καδμίου που εξάγεται για την αποκαδμιοποίηση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μια όσο πιο ολιστική και ρεαλιστική προσέγγιση γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε στενοπούς και παροπίδες και ελπίζω ότι το πακέτο αυτό το οποίο θα δημιουργήσουμε θα είναι αποδεκτό στις διάφορες χώρες, ώστε να καλύψουμε διάφορες πραγματικότητες που θα πρέπει να καλύψουμε εμείς εδώ ακριβώς ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους ε, ενδιαφερόμενους να μπουν στην ενιαία αγορά. Γιατί έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία εργάστηκαν και συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, με άλλου ερευνητικού οργανισμού, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε θα ήταν καλό να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να εισέλθουν δηλαδή σε αυτή την ενιαία αγορά και να το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές που υπάρχουν. Η δουλειά λοιπόν που έχουμε μπροστά μα είναι σημαντική και εύχομαι μετά τη δουλειά του σκηνικού σήμερα να κάνουμε σημαντικό βήμα προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Καρδίνη. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στους σκιώδεις και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ βεβαίως να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για κάποιες από αυτές τις ε, προτάσεις συμβιβασμού που νομίζω αποτελούν και μια πολύ καλή βάση για τη συζήτηση που θα κάνουμε ε, σήμερα το απόγευμα για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε γιατί έχουμε τις 853 τροπολογίες ο οποίος είναι ε, τεράστιος αριθμός για γνωμοδότηση. Είναι θέματα για τα οποία ε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε κοινή λύση και πρέπει να σας πω πως ένα θέμα με το οποίο απασχολούν ε, το ένα τρίτο τροπολογιών είναι τα όρια, ο περιορισμός και τα όρια στο κάδμιο στα φωσφορικά λιπάσματα. Ξέρω πως κάποιοι προσπαθούν να νερώσουν τις ε, ε, προτάσεις. Έχουμε και τα όσα είπε η Κομισιόν για να πάμε από τα 60 μιλιγκράμμ στα 40 μιλιγκράμμ ανά ένα κιλό ε, μετά τα τρία χρόνια και στα Στα 30 μετά από 12 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα θέμα που μας ανησύχησε όλους πολύ ήταν η δυνατότητα που έχουμε να ε, εξολογήσουμε επιστημονικά τις συνέπειες του καδμίου και νομίζω ότι κάποιοι προτιμούν να στηρίξουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας λιπασμάτων, εντάξει, αλλά τα λέει η επιστήμη. Είναι πολύ τοξικό το κάδμιο και υπάρχει μόνος ένας τρόπος να μειώσουμε την έκθεση που έχει σε αυτό το, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Πριν από 15 χρόνια η Επιστημονική Επιτροπή για την Τοξικότητα χονομοδότησε και παρόλο που είχαμε διαφορετικές αξιολογήσεις είπαν πως η χρήση των φωσφορικών λιπασμάτων που έχουν 60 μιλιγκράμμ ε, καδμίου ή πάνω οδηγούν σε σώρευση καδμίου στα περισσότερα ευρωπαϊκά εδάφη και μία υποχρέωση γύρω στα, ο περιορισμός γύρω στα 30 θα μειώσει ε, την έκθεση. Δηλαδή το 60 και πάνω δεν βοηθάει. Μόνο όταν είμαστε στα 30 ή κάτι πιο κάτω μιλιγκράμμ μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτίωση μέσα στα επόμενα 100 έτη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί γιατί εδώ δεν έχει ληφθεί υπόψη ε, και η επιστημονική τεκμηρίωση. Τώρα για το κατά πόσο εμείς εισακούμε τα επιχειρήματα των γεωργών και του γεωργικού κόσμου να σας πω πως έχουμε επενδύσει πάρα πολύ ε, σε τεχνολογία αποκαδμιοποίησης ε, και μέσω της ΕΤΕ και νομίζω ότι αφού έχει απορροφηθεί ε, το κάδμιο από τα φυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε απορρίπανση άρα λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε τους γεωργούς από τα συσσαγωγικά βρώμικα λοιπάσματα εκτός αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε κάδμιο κάτι οποίο θα επηρεάσει και το κατά πόσο μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις εθνικές αγορές και μέσω εθνικής νομοθεσίας, γιατί υπάρχει και εκεί το θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Η νομοθεσία που επιτρέπει τη χρήση του CE θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε πιστεί στην ομάδα μου πως θα πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Δεν θέλουμε τους περιορισμούς που έχει προτείνει η συγγήτρια. Μιλάμε για τα 40 μιλιγκράμμ. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο και θα πρέπει ε, σε 8 χρόνια να προχωρήσουμε και στα 20 μιλιγκράμμ ανά κιλό και να διαδώσουμε τις πληροφορίες που θα επιτρέψει και στους γεωργούς και στους καταναλωτές να μπορούν να γνωρίζουν τι αγοράζουν όταν προμηθεύονται λιπάσματα. Να γνωρίζουν ποιο είναι το περιεχόμενο σε κάδμιο, ε, κυρίως στα λιπάσματα που φέρουν τη σήμανση CE. Αυτά έχω να πω και ελπίζω πως στις επόμενες εβδομάδες και οι θα πετύχουμε στο να βρούμε την κοινή βάση έτσι ώστε να έχουμε ισορροπημένες προτάσεις για την έκθεση αυτή και να μην δαπανίσουμε δύο μέρες ολόκληρες δύο μέρες ολόκληρες γιατί κάθε μία τροπολογία από τους 853 που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Um, πάρα πολύ. Δεν είμαι εγώ ισχύω της εισηγήτρια αντικαθιστώ τον κύριο Νίκολσον. Εμείς στηρίζουμε τα μέτρα για να διαφλεχτεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά η φοιτηρία πρέπει πάντα να είναι τα επιστημονικά στοιχεία και μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Για το κάδμιο υπάρχει μεγάλη συζήτηση από όταν πρότεινε η Κομισιόν τα 60 μιλιγράμμα κιλό μόνο σε αφετηρία, ε, η οποία θα μειωθεί, αλλά είναι προφανέ ότι η Κομισιόν έχει βαστεί σε κάποιε μελέτε οι οποίε εντωμεταξύ έχουν ενημερωθεί 80 μιλιγκράμμ ανά κιλό με την πρόθεση αναθεώρηση θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ασφαλή ε, χρήση, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι έτσι μπορεί να αποφευθεί η συσσόρευση στο έδαφος. Τα 80 μιλιγκράμμ ως μάξιμου σημαίνει ότι ο μέσο όρο θα είναι χαμηλότερο, οπότε θα μειώνονται τα επίπεδα καδμίου γρηγορότερα και θα διαφυλάξουμε έτσι το περιβάλλον χωρίς να επιβάλλουμε υπερβολικό κόστος στους παραγωγούς. Θα εξακολουθεί να είναι μακράν το πιο φιλόδοξο όριο παγκοσμίω. Τα χαμηλότερα όρια επίσης ε, δεν στηρίζονται στα υφιστάμενα επιστημονικά δεδομένα. Ε, άκουσα τον κύριο Πότς. Βεβαίως, δέχομαι όλοι. Δέχονται ότι το κάδμιο είναι βαρύ μεταλλό και πρέπει να το μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά φοβάμαι ότι ακούμε ε, τα συνήθη. Δηλαδή μπερδεύουμε τον κίνδυνο με την έκθεση και μια ακραία θα έλεγα άποψη ότι θα πρέπει τελικά να το μειώσουμε στο 20. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι αυτό ε, σημαίνει οποιαδήποτε περαιτέρω διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Καθόλου και η χρήση της φράσης ε, να νερώσουμε ε, είναι μια υποτιμητική φράση η οποία δεν χρειάζεται. Εμείς μιλάμε για να ορίσουμε ένα επίπεδο το οποίο είναι επιστημονικά συμπεφωνημένο ως το όριο εντός του οποίου μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο και είναι σαφώς εντός των αποδεκτών ε, ορίων. Και εκεί πρέπει να βασιζόμαστε. Ε, εξάλλου μιλάμε για μια ουσία η οποία εμφανίζεται στο περιβάλλον ε, και ποτέ δεν θα εξαλειφθεί πλήρω και έχει συνεπάρξει ο άνθρωπος με αυτήν. Ε, δεν λέμε να το τρώμε κάθε, αλλά παρ' όλα αυτά 80 μιλιγκράμμ είναι ένα επιστημονικά αποδεκτό όριο α, εντός των χωρίων και όπως είπα θα είναι μακράν ο πιο φιλόδοξος στόχος παγκοσμίω. Η αγορά των λοιπασμάτων στην Ευρώπη ήδη έχει μεγάλη συγκέντρωση, δηλαδή πληρώνουν οι καταναλωτές η παραγωγή πολύ υψηλή τιμή και δεν πρέπει να τα ανεβάσουμε ακόμα Λοιπόν, η ε, κυρία Νίκολσον θα ήθελα να ευχαριστήσει ο κύριος Νίκολσον, την κυρία Γκαρντίνη και της εύχεται καλή επιτυχία με τις 800 και πλέον τροπολογίες και καλή τύχη με την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Φέντριλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, είναι τεχνικό και τεχνικό, θα έλεγα. Και βλέπουμε πως υπάρχουν ε, και διαφορετικές κατευθύνσεις. Το είδαμε αυτό και στη συνεδριά των σχεδόν και θα έχουμε και άλλη μία απόψε. Λοιπόν, ανάλογα βεβαίω με την οπτική γωνία του καθενό, ε, βλέπει ο καθένα τα πράγματα διαφορετικά. Η Σουηδία ήταν μία από τι χώρε που ήδη δεκαετία του 1980 είχαν επιβάλει αυστηρά όρια μαζί με την Φιλανδία, την Τσεχία και κάποιε άλλε χώρε, 40 μιλιγκράμμ. Οπότε έχουν ξεπεράσει την πρόταση αυτή ήδη ε, πριν από 30 χρόνια. Και βεβαίως το σκεπτικό ήταν ε, να έχουμε όσο το δυνατόν ε, μικρότερη έκθεση σε μια καρκινογονούσια. Δηλαδή, θα μας επηρεάσει ούτως ή άλλως ό,τι να κάνουμε με την ρήπανση και το κάπνισμα. Επίσης, να δούμε το πού βρισκόμαστε στην έρευνα και το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτή την ομοθεσία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση της ε, Σουηδίας ήθελε να μειώσει το όριο ε, στα 20 μιλιγκράμμα, αλλά το σταμάτησε η Κομισιόν, καθώς δεν υπήρχε στήριξη και ε, δεν υπήρχε κάποια βάση στον κανονισμό. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε παραπέρα να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μιλάμε λοιπόν όχι για μια απαγόρευση. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν θέλει κανείς την πιστοποίηση CE για να μπορεί να εμπορεύεται τα λοιπάσματα αυτά, τότε θα πρέπει να πληρεί κάποιους όρους. Εάν π.χ. πάμε στα 80 μιλιγράμμα, αυτό σημαίνει πως πολλές χώρες οι οποίες έχουν αυστηρότερα κριτήρια θα πρέπει να ε, νερώσουν το δικό του το επίπεδο. Αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν υψηλότερο επίπεδο μπορούν να το έχουν. Αλλά τότε πρέπει να φροντίσετε να κυκλοφορούν μόνο στη δική σας αγορά και να μην τα πουλάτε αλλού. Επίσης υπάρχει και βιολογικά λοιπάσματα που έχουμε συζητήσει και προσπαθήσαμε να βρούμε το νομικό πλαίσιο, πράγματα πολύ ενδιαφέροντα για την κύκλική οικονομία. Έχουμε πολλά φωσφορούχα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και νομίζω ότι αν πετύχουμε αυτό το νομοθέτημα θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τις νέες αγορές, την εγχώρια παραγωγή και ελπίζω να μειώσουμε και τα επίπεδα καρκίνου λόγω έκθεσης στο κάδμιο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα σε τεχνικά και νομικά ζητήματα, αλλά ελπίζω να υπάρξει καλή συνεργασία των σκιωδών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, εκ ε, της ΓΚΟΥ στον κύριο Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Γκαρντίνη. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα Γι' αυτό θα κάνω κάποιες γενικές σκέψεις ως μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ και ως μέλη πρέπει να φροντίσουμε στις ε, συζητήσεις αυτές ε, φροντίσουμε να μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό των ουσιών εκείνων τα οποία βλάπτουν την υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς έτσι περιορίζεται σημαντικά η βιοπικιλότητα. Επίσης, πρόκειται για την υγεία των ίδιων των εδαφών και των μικρότερων μορφών ζωής που υπάρχουν εκεί και ε, συνεισφέρουν στο να μιλάμε για υγιή εδάφη. Θα πρέπει επίσης να δούμε το πώς θα αυξηθεί το ποσοστό οργανικών και μεταλλικών λίπασμάτων τα οποία δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη και στα ύδατα. Και βεβαίως επειδή μιλάμε για κύκλο ο οποίος επηρεάζει και τους αγρότες και τελικά τους καταναλωτές και για να μειώσουμε και την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μικρότερη χρήση τέτοιων βαρέων μετάλλων. Γι' αυτό απαιτείται κατεπηγόντως ε, το κάδμιο, μόλιβδος και ο υδραργύρος να απαγορευτούν και όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο. Νομίζω αυτή είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση. Αυτή ε, είναι η προσέγγιση και κάποιων κρατών μελών που έχουν ήδη απαγορεύσει λοιπάσματα με κάδμιο. Και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση με αυστηρούς ελέγχους και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Το 2003 η Κομισιόν υποσχέθηκε μία πρόταση κανονισμού για το ποσοστό καδμίου στα μεταλλικά λοιπάσματα και χρειάστηκε πολύ καιρό μέχρι να κάνει κάτι, αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Και βεβαίω θα πρέπει και ο νομοθέτης σε συνεργασία με την βιομηχανία να λύσουν το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε προς μία λύση η οποία θα βοηθάει και τον κλάδο να έχει τα κέρδη του χωρίς να βλάπτει την υγεία. Γιατί αν ε, μιλάμε από τη μία για την υγεία και από την άλλη για οικονομικά συμφέροντα, δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε. Αναμένω λοιπόν ε, με αγωνία την απόψινή ε, συνάντηση, αλλά συνολικά θεωρώ ήδη ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσω τώρα το λόγο σε όσους το έχουν ζητήσει. Η κυρία Ρίς είναι η πρώτη μας ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Την πρώτη φορά που κάναμε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό, αν θυμάμαι σωστά το Φεβρουάριο, είχα συνοπτικά παρουσιάσει τα θέματα που εγώ θεωρώ πιο σημαντικά. Καταρχήν πρέπει να υποστηρίξω και εμείς το στόχο της γήτρες και της Επιτροπής, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα οργανικά λοιπάσματα για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία και αυτό σημαίνει βέβαια σταδιακή μείωση των ρηπογόνων ουσιών στα λοιπάσματα. Για τη μείωση λοιπόν των ρηπογόνων αυτών ουσιών το πιο σημαντικό ε, είναι να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές που έχουμε στο θέμα του καδμίου με έναν τρόπο που θα είναι εύχριστος, που θα είναι ρεαλιστικός. Όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν τι τις ίδιες πηγές προμήθειας ε, μέσω εισαγωγών των φωσφορικών λιπασμάτων Όπως επίσης δεν έχουν και την ίδια οξύτητα εδαφών τα κράτη-μέλη λόγω φυσικών συνδικών, όπου καμιά φορά λόγω ακριβώς αυτής της οξύτητας ε, χειροτερεύει η κατάσταση με το κάδμιο στα εδάφη. Εσείς μιλήσατε για τις 853 τροπολογίες. Ε, σας συγχαίρω έτσι και αλλιώς εκ των προτέρων, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολλές, πάνω από 50 έχουν να κάνουν με το κάδμιο. Οπότε νομίζω υπάρχουν αρκετέ γραμμέ ενδεχόμενου συμβιβασμού. Η κυρία Γκροστέτ που δεν είναι εδώ για λόγους που όλοι κατανοούν ε, είχε πει γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουν εκλογές στη Γαλλία είχε πει λοιπόν για τρεις τροπολογίες πρέπει να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση μεταξύ των όσων προτείνει η Συγήτρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μείωση της, ε, της εξάρτησης που έχουμε από την εισαγωγή λιπασμάτων, φωσφορικών λιπασμάτων με μεγάλη κάτια σε κάδμιο και να βάλουμε κατόφλια τα οποία θα είναι φιλόδοξα. Τα 40 μιλιγκράμμ νομίζω μπορούμε να το πετύχουμε και θα πρέπει να πούμε μέσα σε έξι έτη, όχι πιο νωρίς. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο συνάδελφο που πήρε το λόγο πριν από μένα. Θα ήθελα να καταλάβετε Ποια είναι η θέση μας, γιατί μιλήσατε για υποταγή στα λόμπι και στου παραγωγούς. Όχι, εγώ είπα πριν από κάποιους μήνες πως θα πρέπει να δούμε και την σκοπιμότητα και το κόστος και το κατά πόσο είναι ε, δυνατόν με πρακτικό τρόπο να εφαρμοστούν όλα αυτά και νομίζω ότι τότε μας είχε κάνει και μια παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας είχε πει ότι μέχρι στιγμής οι τεχνικές που θα επιτρέψουν να πετύχουμε αυτά τα κατόφλια δεν είναι ακόμα διαθέσιμα διαθέσιμες. Οπότε, ναι, ας στοιχηματίσουμε αυτών στο μέλλον, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά με τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κραδένουμε τώρα το λάβαρο του υποταγή στα λόμπι. Για την 430 ε, τροπολογία να σας πω που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο τα νέα όρια που προτείνονται ε, μπορούν να επιτευχθούν. Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες. Και εδώ έχουμε την τροπολογία επίσης 421 που μιλάμε για τα χαμηλότερα κατόφλια που είναι 20 μιλιγκράμμα ανά κιλό και για την σήμανση που θα περιγράφει τα όρια. Πολύ ρεαλιστικό, πολύ σωστό. Πρέπει οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα λοιπάσματα και έχουμε και την 773 που ζητά να έχουμε και ενδείξεις ε, για τα βαρέα μέταλλα σε όλα τα λοιπάσματα που φέρουν τη σήμανση CE. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν δηλώνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλο. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να το κάνουν έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον, η ανθρώπινη υγεία και για παράδειγμα να ενημερώνουμε και να ε, επικαιροποιούμε σχέδια δράσης σχετικά. Ένα τελευταίο σημείο, να μιλήσω για τα θέματα που έθεσε η συγγήτρια και που θεωρώ πιο σημαντικά. Για την νέα νομοθεσία νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα υποπροϊόντα και τα κατάλοιπα και άλλα απόβλητα έτσι ώστε η κυκλική οικονομία να λειτουργήσει καλύτερα και νομίζω η δεύτερη γραμμή συμβιβασμού θα πρέπει να είναι για τα υπόλοιπα απόβλητα που ε, ανακτώνται. Ζητά η κυρία Καρδίνη ο κατάλογος αυτός να επεκταθεί και θα τη στηρίξω βεβαίως στο αίτημά αυτό, που είναι η δεύτερη γραμμή από τις οποίες θα μπορούσαμε εμείς να συμβιβαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγιούσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως έχουμε ένα σημείο συμφόρησης με τη συγκεκριμένη νομοθεσία και το σημείο συμφόρησης εδώ ακριβώς είναι το κάδμιο. Τα όρια που ορίζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα, την περιβαλλοντική τοξικότητα και το περιβάλλον που ζήτησαν τα όρια αυτά να βασίζονται σε μια έκθεση αξιολόγησης κινδύνου. Και το 2015 η Επιτροπή αυτή μας είπε πως δεν έχουμε σόρευση στα εδάφη, γιατί αν παραμείνουμε κάτω από τα 80 ε, μιλιγκράμμ ανά χιλιόγραμμο. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μόνο τι κάνουν η Σουηδία, η Αυστρία και η Φιλανδία. Είναι χώρες που έχουν μικρή γεωργική παραγωγή, που έχουν χαμηλή χρήση λιπασμάτων και που έχουν ε, πετρώματα με μικρή περιεκτικότητα σε κάδμιο, σε κοιτάσματα πολύ κοντά τους. Ας δούμε όμως τι κάνουν οι υπόλοιποι. Η νομοθεσία αυτή δεν λαμβάνει υπόψη πως έχουμε διαφορετικά εδάφη στις διαφορετικές περιφέρειες. Στη χώρα μου, στην Ισπανία η απορρόφηση του καδμίου είναι πολύ μικρότερη από ό,τι σε χώρες με πιο υγρά κλίματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει μια διαδικασία αποκαδμιοποίησης από τα φωσφορικά ε, πετρώματα στις χώρες προμηθευτές. Μα αυτό δεν είναι σε βιομηχανικό επίπεδο σήμερα βιώσιμο. Οι τροπολογίες μας λοιπόν από την Ισπανική Αντιπροσωπεία στο ΕΛΚ είπε πως θα πρέπει να είμαστε στο 45 ε, μιλιγκράμμα ένα κιλό και είμαστε κατά οποιασδήποτε μείωσης κατά από τα 75, εάν δεν εμφανιστούν κάποιες βιομηχανικές επεξεργασίες που θα επιτρέψουν μια πιο εύκολη αποκαδμιοποίηση αυτών των πετρωμάτων. Έχουμε τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και ένα νέο εκτιμώντας όπου είπαμε πως το πέτρωμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί πρώτη ύλη ζωτικής σημασίας, δηλαδή όπου υπάρχει περίπτωση να σπανίσει η προμήθεια ή ένα νέο άρθρο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει σε πέντε χρόνια μετά τη θέση εφαρμογή του κανονισμού μια έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτού και για το κατά πόσο έχει μειωθεί ε, το ποσοστό ρήπανσης. Αυτά να τα λάβετε υπόψη εσείς οι εισηγητές γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και όπως είπα και εγώ έχουν ληφθεί υπόψη οι αξίες χωρών που έχουν νομοθεσία σύμφωνα με τα όσα οι ίδιες χρησιμοποιούν, καταναλώνουν και χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδελφοί. Η κυρία Πριστά Εξώματος Επιτροπής. Thank you very much, Chair. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σημαντικός ο φάκελος αυτός, υπόθηκε κιόλας, ά τα πρώτα παραδοτέα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης και κλικής οικονομίας και συμφωνώ με αυτό υπόθηκε ότι είναι περίπλοκο ζήτημα και νομικά και τεχνικά. Δηλαδή, εδώ διασταυρώνονται διάφορες νομοθεσίες για τα, για τα απόβλητα, τα απορρίμματα, χημικές ουσίες κλπ. Και πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση πριν ληφθούν θέσεις. Οπότε θα σας δώσω μόνο τη δική μας προκατακτική ανάλυση. Εμείς θεωρούμε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά σε αυτό τον φάκελο με αυτές τις τροπολογίες και θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από αυτές, τις νέες, τις καινούργιες που είδαμε τώρα. Έχουμε τη θέσπιση νέας ορολογίας σε κάποιες τροπολογίες. Αντί για ανόργανα λέμε ορυκτά λοιπάσματα ας πούμε. Κάνουμε διάκριση μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών ε, θρεπτικών ουσιών και άλλα παραδείγματα. Θα μπορούσα να πω σε γενικέ γραμμές ότι θα εξετάσουμε θετικά τις τροπολογίες που ακολουθούν την τρέχουσα ορολογία ώστε να αποφευθεί βέβαια και σύγχυση. Και επίσης συμμεριζόμαστε τις απόψεις της εισηγήτριας και άλλων ότι αυτός ο κανονισμός θα ενισχύσει τι επενδύσει στην κυκλική οικονομία και στόχος μα εμάς ως Κομισιόν εδώ είναι η ανάκτηση και γι' αυτό ακριβώς θα εξετάσουμε θετικά τις τροπολογίες που θα αξιοποιούν ακριβώ την ανάκτηση στα πλαίσια της κυκλική οικονομίας. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο να τονίσω έτσι έξι αρχικές μας ανησυχίες. Ε, πρώτη αφορά τα, τους βιοδιογέρτες, φυτών. Θεωρούμε ότι η γραμμή που χωρίζει αυτό το σημείο με την τρόξα νομοθεσία πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Γιατί θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι γίνεται με τα λοιπάσματα που έχουν τη σήμανση της Ένωσης. Και μία από τι ανησυχίε μας είναι η πρόταση για περίπτωση προϊόντων που ενισχύουν τη βιωτική αντοχή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα προϊόντα δεν χρειάζεται απαραίτητα να εξαφανιστούν από την αγορά, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται υπό την τρόσα νομοθεσία για τα φυτά, για τα φυτικά προϊόντα. Μετά, είδαμε τα παράγωγα, τα παράγωγα προϊόντα, ζωτικά παράγωγα, σε κάποιες τροπολογίες. Οπότε καταλάβαμε λένε κάποιες τροπολογίες ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται εδώ η σήμανση, πρέπει να εφαρμόσετε τη σήμανση, έστω και να λείπουν κάποια στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παράγωγα θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα λοιπάσματα με σήμανση ε, ε, χωρίς καμιά διαδικασία απολύμανσης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει ένας κίνδυνος Μεγάλο κίνδυνο για την υγεία και για το περιβάλλον, κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Τρίτον, εξετάσαμε κάποιες τροπολογίες που αφορούν το REACH και την καταγραφή, ιδιαίτερα τις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις χημικού κινδύνου. Μέχρι τώρα, αυτές οι αξιολογήσεις είναι απαραίτητε για όλες τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα χημικά προϊόντα, έστω και βρίσκονται σε χαμηλή περιεκτικότητα. Γιατί είναι ο μοναδικό κίνδυνο αξιολόγηση που απαιτείται για τι πρωτογενεί χημικέ ουσίε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτέ τι ε, προποθέσει ακριβώ καταγραφή του ρίτς, έστω και με χαμηλή περιεκτικότητα. Αν αφαιρεθεί αυτό, θα έχουμε κινδύνου ανυπολόγιστου και θα είναι δύσκολο να του ελέγξουμε. Τέταρτη παρατήρηση σε αυτή τη φάση. Τα ορυκτά λοιπάσματα. Υπάρχουν προτάσεις για περιορισμό των προϊόντων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ορυκτά λοιπάσματα. Ιδιαίτερα το 1% ας πούμε ορυκτού οργανικού συγγνωμιά, άρθρακα ε, και μετά τα φωσφορικά αλάτα. Θεωρώ όμως ότι κάνοντας αυτό αποκλίνουμε πολλά από τα καινοτόμα θρεπτικά συστατικά, ανάκτησης μάλιστα, που θέλουμε να περιληφθούν. Και για άλλα καινοτόμα προϊόντα ισχύει το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει εμφανής λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ούτως ή άλλως οι γεωργοί θα πρέπει να ενημερώνονται σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, σε σχέση με την ε, διαλυσιμότητα των φωσφορικών αλάτων μέσω της σήμανσης. Και τώρα που εξετάζουμε κανόνες ανάκτησης για προϊόντα στάχτης και άλλα, εξετάζουμε και άλλα κριτήρια αγρονομικά, υγειοπονικά, τα οποία θα προτείνει η Κομισιόν στο μέλλον να υιοθετηθούν. Οπότε διατρέχουμε ένα κίνδυνο εδώ όσον αφορά τη σήμανση και την ενημέρωση του Γεωργού. Ένα πέμπτο σημείο αφορά τα νητρικά και την οδηγία. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ καθορίζουμε κανόνες ε, που αποτρέπουν την ε, μόλυνση των υδάτων και δεν περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες την λιματολάσπη και τη χρήση της σε κάποιες περιοχές. Όμως υπάρχουν τρόποι παρέκκλησης από αυτό το όριο αν τεκμηριώνεται ε, περιβαλλοντικά και γεωπονικά. Η Κομισιόν πρότεινε αυτό τον κανονισμό χωρίς τροπολογίες για τα μητρικά και η τροπολογίες νομίζω εδώ δεν σχετίζονται με αυτές τις ε, οδηγίες για τα αντιτρικά. Έχουμε δύο διαφορετικές λοιπόν νομοθεσίες, κανονισμός και οδηγία. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά πεδία εφαρμογή και διαφορετικοί στόχοι. Οπότε θεωρούμε ότι εδώ αυτά πρέπει να εφαρμοστούν συμπληρωματικά. Οπότε δεν συμφωνούμε με τις τροπολογίες που αφορούν τα νητρικά. Τέλος, για το κάθμιο δύο λόγια. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για διάφορες τροπολογίε. Δεν είναι μυστικό ότι η Κομισιόν διστάζει να μειώσει τους φιλοδοξού στόχους για το κάδμιο. Αντιπροτείνεται εδώ πέρα σε κάποιες περιπτώσει μία ρήτρα ανθεώρησης για τα υψηλά όρια. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο status quo γιατί στην, οι επενδύσεις αποκατημοποίησης δεν θα γίνουν διαφορετικά και μια ρήτρα αναθεώρησης απλά και μόνο θα λέει δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν δεν συνοδεύεται δηλαδή από πολύ φιλόδοξους που θα πρέπει να τεθούν από τώρα. Από πολύ φιλόδοξες αξίες. Τώρα, για τα φωσφορικά άλατα και κατά πόσο θα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο με τα κατάργαστα υλικά. Νομίζω αυτό δεν είναι σωστό. Εξάλλου έχει αναφερθεί εδώ και επανειλημμένος ότι 80 μιλιγκράμμ ανά κιλό ότι ενδεχομένως είναι ασφαλές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. 80 λοιπόν μιλιγράμμα ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτηση και το 2013 θεωρούσαμε ότι ήταν το όριο μη συσσόρευσης. Υπάρχουν όμως δύο λόγοι εδώ για τους οποίους η μη συσσόρευση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές επίπεδο. Καταρχάς, υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα σε σχέση με το επίπεδο μη ε, συσσόρευσης σε διάφορε χρονικές στιγμές. Ας πούμε το 2000, στις αρχές του 2000, θεωρούσαμε ότι ήταν τα 20 μιλιγράμμ. Το 13 ας πούμε θεωρούσαμε ότι ήταν τα 80 μιλιγκράμμ ανά κιλό πράγματι. Όμως στην αρχή του τρέχοντος ε, είχαμε πει ότι ήταν 70. Υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα σε σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία. Και πάλι μιλάμε για επίπεδο μη συσσόρευσης. Δηλαδή το επίπεδο στο οποίο η ρήπανση, η τρέχουσα ρήπανση παραμένει σταθερή. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να πούμε ότι δεν υπάρχει σαφές όριο. Γιατί το status quo στην ρήπανση δεν σημαίνει ότι η έκθεση στο κάδμιο είναι ασφαλής. Και αυτό είναι και ξεκαθαρό αν δείτε τις μελέτες της ε, ΕΦΣΑ σε σχέση με τις εκθέσεις. Τις διατροφικές που λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί η διατροφική έκθεση επειδή ακριβώς ε, το κάδμιο θέτει κίνδυνο στην ανθρώπινη αγία κλπ. κλπ. Δύο λόγια να σας πω επίσης για τις προτάσεις για θέσπιση αυστηρότερων ορίων. Θεωρούμε τώρα ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό της αγοράς και όσο πιο μεγάλη και επαρταμένη περίοδος περισσότερο κατακαιρματισμό θα οδηγήσει. Και αυτός είναι από τους κύριους στόχους εδώ, δηλαδή το να ανοίξει η αγορά για τα λοιπάσματα. Κάτω το οποίο γίνει αυτό θα χαθεί ο στόχος. Καταλήγω λοιπόν. Αυτά είναι κάποια από τα προκατακτικά μας σχόλια. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές των τροπολογιών που ξέρω θα αναλύσετε και θα συζητήσετε τους ερχόμενους μήνες και από τη δικιά μας πλευρά και εγώ και οι συνάδελφοι είμαστε έτοιμοι πραγματικά να σας βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μας. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση αυτή που αποδεικνύει το ότι υπάρχει πραγματικά ένα βρασμός για διάφορα σημεία. Και αυτό είναι καλό γιατί νομίζω ότι με δίνει μια ζωντανή εικόνα. Εγώ επανέρχομαι στο αρχικό μου το κριτήριο, δηλαδή εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε κυρίως να υποφεληθούμε από την εμπειρία που υπάρχει και που είδαμε από τις παραβάσεις των σαντέλφων στις διάφορες χώρες και που σχετίζεται αυτή η εμπειρία με την πραγματικότητα Ξεκινώντας από τα εδάφη, όπως ο Λεγισνάδελφος Δρύς, ας πούμε. Είναι προφανές ότι η μικρή Σουηδία, η οποία έχει, ας πούμε, ορυκτά με πολύ χαμηλό επίπεδο υπεριοκτακαδμίου κοντά στη Ρωσία ας πούμε, και, λοιπά, και, περιορισμένη η παραγωγή έχει διαφορετική άποψη από χώρες ας πούμε, οι οποίες έχουν μια γεωργία πολύ πιο μαζική και με δάφη τελείω ε, διαφορετική φύση και με τελείω διαφορετικέ εισαγωγέ. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η εμπειρία τη Ιταλία εδώ είναι εμπειρία θεωρώ πολύ θετική γιατί είναι μια χώρα που έχει μια πολύ ισχυρή γεωρική συνιστόσα έχει και πολύ χαμηλά επίπεδα το είπε και η Κομισιόν από τη στιγμή που τέλο πάντων δεν υπάρχουν ξεκάθαρα όρια για το κάδμιο. Εμεί οπωσδήποτε βέβαια θα βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Απλά και μόνο δηλαδή θέτοντα ένα συγκεκριμένο όριο, γιατί τα διάφορα όρια που ακούσαμε είναι όρια που είναι το ίμιση του πιο αυστηρού που ισχύει παγκοσμίω. Αν κοιτάξουμε χώρες αξιόλογες, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, όπου υπάρχει τέλο πάντων φροντίδα για το περιβάλλον και ευαισθησία. Η Ιταλία λοιπόν αναφέρθηκε πρόσφατα ως η πιο υγιής χώρα στον κόσμο. The healthiest, λέει η ομιλήτρια. Οπότε νομίζω εδώ αυτό προσφέρει και κάποια αξιοπιστία, έτσι δεν είναι. Επειδή είναι μια χώρα η οποία ανέκαθεν επέδειξε μεγάλη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Οπότε εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι πάρουσε εμπειρίε, επειδή αν ξεκινήσουμε μόνο από τη θεωρία, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να αποκλείσουμε, να κάνουμε δηλαδή αποκλεισμού και αντί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για όλου, να αν πάμε πολύ μακριά, αν βάλουμε ξέρω εγώ 20 μιλιγράμμα ένα κιλό μεθαύριο, το λέω παράδειγμα έτσι, παράδειγμα μη ρεαλιστικό, αλλά τέλο πάντων είμαστε έτσι πολύ βολονταριστέ και διατρέχουμε, διατρέχουμε τον κίνδυνο μάλλον να πετύχουμε το αντίθετο. Να κάνουμε κάτι δηλαδή το οποίο θα αφορά λίγου και θα ισχύσει τελικά. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Λαμβάνοντα υπόψη την πραγματικότητα. Να βρούμε κάτι λοιπόν και εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό εις όφελος όλων των ε, πολιτών. Αλλιώ θα κάνουμε κάτι το ελιτιστικό υπάρα αυτών δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν πολλά και για τα βιολογικά, γιατί και τα βιολογικά πούμε, στις διάφορες χώρες ε, είναι για τους έχοντες και τους κατέχοντες που μπορούν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα για να φάνε βιολογικά ας πούμε. Ποιος τρώει βιολογικά σε καθημερινή βάση ας πούμε, στη χάση και στη φέξε σε κάποιες χώρες. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα που να μην είναι για λίγους και να είναι καλά δηλαδή για λίγους και λιγότερα καλά για τους περισσότερους. Αυτό εγώ θεωρώ σημείο ισορροπίας που θα πρέπει να αναζητήσουμε σε όλα τα παιδιά, έτσι. Να πάντως υπόψη, ξαναλέω τις διάφορες πραγματικότητες που ισχύει που ισχύουν ας πούμε στην Ολλανδία, στη Σουηδία κτλ. Σε όλες τις χώρες διαπρέπουμε σε κάτι. Ας τα λάβουμε λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά για να καταλήξουμε σε κάτι καλό για τα εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων που προσβλέπουν σε εμά για κάτι το οποίο θα τους προστατεύει στην υγεία τους, όχι όμως για κάτι υπερβολικό που θα αφορά λίγους Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ στις 30 Μαΐου, στην ΙΜΚΟ στις 13 Ιουλίου και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 17. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι τελείωσε η ημερήσια διάταξη για την πρώτη αυτή συνεδρία της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Σας δίνω λοιπόν ραντεβού να τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.